Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση γιατί περνάει και ο χρόνο. Ελπίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα έλθουν εγκαίρω τουλάχιστον πριν την ψηφοφορία. Ξεκινήσουμε με το σημείο 10 τη ημερησία διάταξη. Από εκεί που είχαμε μείνει το πρωί. Μαρή Τερέζα Σμιθ. Ε, έχουμε τι προκλήσει για την εδαφική συνεργασία, τη μελλοντική ατζέντα για τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Στόχος 3. Να δώσω το λόγο στη Μαρή Τερέζ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη ε, που μα επιτρέπει σήμερα να έχουμε αυτή την αντιλογή απόψεων για την Ευρωπαϊκή Διαπεριφερειακή Συνεργασία. Είμαι σίγουρη ότι η συζήτηση που έχουμε σήμερα το απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα πλούσια και θα μα επιτρέπει να εμπλουτίσουμε και τον προβληματισμό μα. Επίση, ε, ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή Σαρλ Ρίκ και τον κύριο Μαρτίν Κουρανιάη που είχαν την ε, ευγενική ε, καλοσύνη να δεχτούν ε, την πρόσκλησή μας και να κάνουν το ταξίδι και μέχρι εδώ, γιατί δεν ήταν κάτι προφανές λόγω και του καιρού σήμερα και ε, είναι και οι δύο εμπειρογνώμονες ε, για την ενταφική συνεργασία στην Ευρώπη. Ο καθηγητή Σαρλ Ρίκ ε, το συνάντησα σε μια διάσκεψη για τις πόλεις στην Επιτροπή των Περιφερειών και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης στο Περιτήριο Ευρωπαϊκών Περιφερειών τα ακαδημαϊκά, τα ακαδημαϊκά έργου που έχουν συνταχθεί για το Σύνολο της Ευρώπης και για το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι σε μια αναφορά για κάθε δεσυνοριακό παράγοντα. Αναφέρομαι κυρίω στο χειρίδιο δεσυνοριακή συνεργασία, το οποίο δημοσιεύτηκε πολλάκι και δεν μεταφράστηκε σε πολλέ γλώσσε. Ο κύριο Μαρτίν Κιγέρμο Ραμίζρε είναι γενικό γραμματέα τη Ένωση ε, Παραμεθαρίων Ευρωπαϊκών Περιφερειών ε, γιατρό, ε, κατα... εργάζεται σήμερα στο πλαίσιο τη Ένωση Παραμεθαρίων Ευρωπαϊκών Περιφερειών η οποία ιδρύθηκε το 71 και είναι η πιο αρχαία, η πιο παλιά ε, Ένωση. Ο συνάδελφος Βένιστεν Ρο ήταν ο πρόεδρος ε, από το 2004 στο 2005 αυτής της Ένωσης. Στις 28 Οκτωβρίου στην περασμένη συνεδρίαση κάναμε για πρώτη φορά μία πρώτη συζήτηση με πλούσια ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον του στόχου 3. Για να σας υπενθυμίσω, η εδαφική ε, ευρωπαϊκή διαπεριφερειακή συνεργασία έχει γίνει το στόχος 3 της πολιτικής συνοχής με 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2003 σαν ε, ε, προϋπολογισμό. Ε, έχουμε τρεις πτυχές, διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεθνική και θέλει να καλύψει τις κοινέ προκλήσεις των περιφερειών. Πολλοί εξημών υπογράμμισαν την προφανή προστιθέμενη αξία της εδαφικής συνεργασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αναγκαιότητα να θέσουμε τους πολίτες στην καρδιά των πρωτοβουλειών μας καθώς ε, εδώ μιλάμε για ε, μια ζωντανή ε, εδαφική και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση το να προωθήσουμε στο πλαίσιο του στόχου 3 το είδος του Εράσμου στον των εκλεγμένων της τοπικής αυτοδιοίκησης έτυχε επιτυχίας. Ε, η χρηματοδότηση βέβαια του στόχου 3 πρέπει να αποσαφινιστεί. Εγώ νομίζω ότι η μακροπεριφερειακή λογική θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ευέλικτη τη εδαφική συνοχή έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσαρμοστεί και να αποφεληθεί τα μάλλα. Από την τελευταία συζήτηση που είχαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημεσίευσε την πέμπτη έκθεση για την πολιτική συνοχή την οποία χαιρέτησε η Επιτροπή μας ως μια καλή βάση εργασίας. Η έκθεση αυτή ε, στοχεύει σε μια στενή συνδέση μεταξύ πολιτικής συνοχής και στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 χάρη σε μια καλύτερη στόχευση των πόρων και με έμφαση στα αποτελέσματα. Η διάσταση της εδαφικής συνοχής είναι παρούσα ακόμη και αν τα διασυνοριακά ζητήματα ίσως κατά την άποψή μου θα έπρεπε να τονιστούν περισσότερο. Πέρα από το αστικά ζητήματα. Οι προτάσεις τη έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσε σε ό,τι αφορά την ε, οργάνωση περιφερειακών προγραμμάτων ε, και μπορούν ε, να ανοίξουν την οδό για πιο επιχειρησιακά, πολυπεριφερειακά προγράμματα με κοινέ θεματικές. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια ενισχυμένη ε, διαπεριφερειακή πτυχή για τις μακροπεριφέρειες. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα γιατί ε, επιτρέπεται έτσι να έχουμε καλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διάφορων στόχων σε διευρυμένη εδαφική βάση, αλλά η ενίσχυση δεν πρέπει να γίνει βάρος των άλλων πτυχών. Τα συμπεράσματα της άτυπης συνεδρίασης των Υπουργών ε, που είναι αρμόδια για την πολιτική συνοχή που, θα λάβει χώρα, που έλαβε χώρα στη ΛΕΑ 22 και 23 Νοεμβρίου ε, είναι ενθαρρυντικά. Υπάρχει μια συνένεση των Υπουργών για τη διαχείριση τη αρχιτεκτονική του στόχου 3 και κυρίω για την αναγκαιότητα ενίσχυση του στόχου αυτού. Έτσι, αρχίζουμε να βλέπουμε σαφέστερα τι θέσει του καθένα και αυτό θα μα επιτρέψει να φτάσουμε σε μια επικοδομητική και ρεαλιστική θέση του Κοινοβουλίου. Σας ε, ανέφερα τις σκέψεις μου, τώρα θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας που δεν μπορούν να μας δώσουν ε, νέες απόψεις και μια νέα σκοπιά και να μας δώσουν κάποιο προσανατολισμό στη σκέψη μας. Ευχαριστώ την κυρία Σμίθ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρτιν και Γέρμο Ραμύρες. Hello. Yes. Eh, bien, hablaré en español, ya que... Να μιλήσω ισπανικά Καθώ μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και δεν είναι πάρα πολύ συχνό, να μπορώ να μιλήσω στη μητρική μου. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Σάντσε Σμιθ ε, για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μας, γιατί η κύρια δραστηριότητα της Ένωσής μας είναι να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των παραπευθερίων περιοφοριών και εδώ θέλουμε να βρούμε μια σειρά στρατηγικών συμμάχων. Πάντοτε μας χρειάζονται και εμείς εν τέλει Έχουμε πάρα πολύ λίγες δυνατότητες να επηρεάσουμε θεσμούς ε, που πιστεύουν στις πτυχές ε, και σε όσα εμείς ε, υπερασπίζουμε. Εδώ αναφερόμαστε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και έτσι λοιπόν είναι καλό που ερχόμαστε εδώ να υπερασπίσουμε τη θέση μας γιατί κατανοούμε ότι στα κύρια χαρακτηριστικά των πολιτικών που προσδορίζονται εδώ συμφωνούμε απόλυτα έτσι λοιπόν μιλάμε αφενός για επικουρικότητα, για να εντάξουμε την ε, ε, περισσότερο ε, την τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουμε περισσότερη Ευρώπη και από την άλλη και τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στο αυτό να δημιουργήσουμε περισσότερη Ευρώπη. Αυτό είναι ένα ζήτημα γιατί ένα είναι να μιλούμε θεωρητικά, αλλά όταν μιλάμε για πολιτικές και μάλιστα πολιτικέ όπου έχουμε χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, τότε έχουμε διαλεκτική μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού και τοπικού επίπεδου. Και το εδαφικό ζήτημα ή το ζήτημα τη εδαφική συνεργασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Έτσι λοιπόν, εμεί ε, έχουμε ε, εδώ ευρία επιχειρήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα σα εκθέσω όλα. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά τηλεγραφικό και να σα πω ποια είναι τα κυρία σημεία που μα ανησυχούν για το θέμα τη εδαφική συνεργασία, πώ βλέπουμε το μέλλον ποια εντύπωση μας δημιουργήθηκε από το έγγραφο που εκπονήθηκε από την ε, κυρία Σάντσε Σμιθ και να δούμε και ποια είναι ο σχετισμός με τη συζήτηση που γίνεται στα πλαίσια της Επιτροπής των Περιφερειών. Καταρχήν, εμείς ε, είμαστε μια ένωση υπέρ της Ευρώπης. Ε, οι παραμεθόριες περιοχές ε, συμμετέχουν στην ένωσή μας. Είναι απομακρυσμένες από τα κέντρα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, μάλιστα και από τα κέντρα των δύο των χωρών και υπάρχει έλλειψη σημαντική στις υποδομές και οι νέοι όταν έχουν την ευκαιρία φεύγουν ε, σε μια τέτοια τυπική παραμεθόριο περιοχή ένα νέο όταν μπορεί να βρει ένα εράσμου ή ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα που να του επιτρέπει να φύγει, φεύγει. Παρ' όλα αυτά οι περιφερειακέ κυβερνήσεις και εμείς η ίδια η Ένωση προσπαθούμε να καταστήσουμε ελκυστικές τις περιοχές αυτές για να μην φεύγει ο κόσμος. Ε, ε, έχουμε, αν φεύγουν και οι πιο δυναμικοί τομείς της επιχειρηματικότητας δεν έχουμε τίποτα. Έτσι προσπαθούμε λοιπόν να διατηρήσουμε αφήσουμε τους νέους αυτές τις ε, παρενθώρες περιοχές καθιστώντας τις πιο ελκυστικές. Το, ε, ε, πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη τη στιγμή που εκπονούν τι στρατηγικέ ανάπτυξη να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη αυτέ τι παραμεθόριε περιοχέ, αλλά να προσπαθήσουν και να ε, προβούν και σε ένα συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Εδώ μιλάμε για τη διασυνορική συνεργασία και από τα ευρωπαϊκά όργανα αυτό προωθείται εδώ και αρκετέ δεκαετίε. Αυτό αποτέλεσε το θεμέλιο ενό προγράμματο, του προγράμματο Interreg, ιδιαίτερα επιτυχέ, το οποίο ξεκίνησε περίπου πριν 20 χρόνια με λίγου πόρου, προωθώντας ε, σχέδια μικρά peer-to-peer και σήμερα έχει κάπως ε, μεγαλύτερη η χρηματοδότηση. Βέβαια, μιλάμε για γελία πως αν το συσχετίσουμε με το γενικό περιπολογισμό της Ένωσης, όμως ε, ο στόχος είναι πολύ σχετικό και έχουμε συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη και επίσης είναι πολυεθνικά τα προγράμματα, δηλαδή στι διασυνορικές στρατηγικές συνεργασίες θέλουμε να εγγυηθούμε ότι θα εφαρμόζονται κάποια προγράμματα συγκεκριμένα για την ανάπτυξη. Αν δούμε τώρα τι αξιολογήσει που έγιναν για τα τρία στάδια του Interreg, ε, μιλάμε για μια επιτυχία, η διασυνοριακή συνεργασία και αναφέρομαι κυρίω στη διασυνοριακή συνεργασία γιατί είναι το πεδίο που εργαζόμαστε και γιατί σήμερα έχουμε το 75% του συνόλου του εδαφικού στόχου, αλλά το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τη διαπεριφερειακή, για τη διεθνική συνεργασία Δηλαδή, οι περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να δημιουργήσουν δίκτυα ενδιαφέροντος, μπορούν να συντονιστούν και να συνεργαστούν για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους και κανείς δεν είναι κατά αυτού. Αναφερόμουν στις ε, παραμεθόριες περιοχές με τις ιδιαιτερότητές τους, μόνο μέσω το συντονισμό πολιτικών, μέσω των συνόρων και με μια εποπτεία από τα ευρωπαϊκά όργανα είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη για αυτές τις περιοχές. Πέραν αυτού, οι ευρωπαϊκές παραμεθόριες περιοχές όπου υλο πραγματοποιείται μια συνεργασία που να πηγαίνει πέρα από τα προγράμματα και μιλάμε για 50 έτη από τότε που δημιουργήθηκε η πρώτη δομή τέτοια συνεργασία. Είναι πραγματικά εργαστήρια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι πολίτε που ζουν σε παραμεθόριε περιοχέ, όταν υπάρχουν προγράμματα που υλοποιούνται κατάλληλα γνωρίζουν και συνειδητοποιούν πολύ περισσότερο το ευρωπαϊκή διαδικασία οικοδόμησης από πολλούς πολίτε που ζουν στι διάφορε πρωτεύουσε, που για αυτού το ευρωπαϊκό ζήτημα είναι κάπω πιο μακρινό. Για του πολίτε των παραμεθόριων ε, περιοχών ορισμένα από τα προγράμματα που σχεδιάζονται εδώ στι Βρυξέλλε, είναι η καθημερινότητά του, είναι η εγγύηση ότι μπορεί να έχουν το ίδιο επίπεδο ιατρική περιθαλψη ότι υπάρχουν ενεργητικέ πολιτικέ για την απασχόληση ε, για τους παραμεθόριους εργαζομένου. Και τελικά, είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες των παραμεθόριων περιοχών και ε, αυτό μετριάστηκαν ακριβώς λόγω της αποτελεσματικής εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με τον ίδιο τρόπο, επίσης θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκές παραμεθορές περιοχές είναι πραγματικά εργαστήρια της διακυβέρνησης σε πολλαπλά επίπεδα τα τελευταία έτη και κυρίως το τελευταίο έτος ε, έγινε μια σημαντική συζήτηση για το πόσο ε, σκόπιμη είναι αυτή η πολυεπίπεδη κυβέρνηση, για το πώς θα ε, διαχειριστούμε και πώς θα διακυβερνήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επίπεδα έτη. Έτσι λοιπόν αυτή η διαδικασία διακυβέρνηση κρατάει εδώ και 50 χρόνια. Και αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο από τις αντικειμενικές αξιολογήσεις, υπάρχουν και πιο άτυπες αξιολογήσεις, είναι πολύ θετικό. Έτσι σήμερα έχουμε μία εμπειρία τεράστια η οποία μας επιτρέπει να πούμε ότι η χρήση της επικουρικότητας και των διαρθρωτικών ταμείων και των, του Τομείου Συνοχής για να πετύχουμε πιο αποτελεσματική εδαφική συνεργασία ε, αυτό που θα καταλήξουμε, στο οποίο θα καταλήξουμε στο εξή είναι να έχουμε περισσότερη Ευρώπη και να δώσουμε μία νέα δυναμική σε αυτές τις περιοχές. Έτσι λοιπόν τελικά αποκτήσαμε με ένα νομικό μέσο που για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε όλο σε όλη την επικράτεια των Ευρωπαϊκών Μελοδαφικής Συνεργασίας. Αυτό το σε μια συγκεκριμένη στιγμή το 2006 όταν δημοσιεύτηκε, ας πούμε ότι έγινε της μόδας. Τότε διατρέχαμε τον κίνδυνο να μετατρέψουμε όλες τις δομές ε, που παραδοσιακά ασχολούνταν με την εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη, να τους μετατρέψουμε σε τέτοιους ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας. Όμως ε, είχαμε και ικανοποιητικά μοντέλα. Ε, ο Ευρωπαϊκός Ομίλος Εδαφικής Συνεργασίας δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά είναι ένα ακόμη στοιχείο που στα πλαίσια του δημοσίου δικαίου μας επέτρεψε να αρχίσουμε αυτή τη διασυνορική συνεργασία σε τοποθεσίε όπου ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί εδώ ή τώρα είναι πολύ δύσκολο να σα εξηγήσω του λόγου, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι είχαμε διάφορα νομοθετικά διοικητικά συστήματα και διάφορε νοοτροπίε και φιλοσοφίε ε, μεταξύ των συνόρων. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέσο δημοσίου δικαίου που να επιτρέπει την εναρμόνιση τη εργασία σε αυτά τα επίπεδα. Και ε, Κατόπιν των ε, ΕΟΕΣ, των Ευρωπαϊκών Ομήλων, θέλω να αφαιρθώ στι μακρόπεριοχέ. Η νέα μόδα που προέκυψε μετά του ΕΟΕΣ ήταν αυτή η μόδα των μακροπεριοχών. Και επιτρέψτε μου να την αποκαλώ μόδα. Δηλαδή, ε, στι ε, περιοχέ αυτέ δημιουργήθηκε μία κοινότητα εργασία, κατόπιν ένα Ευρωπαϊκό ομω Εδαφική Εργασία και τώρα θέλουν να δημιουργήσουν μία μακροπεριφέρεια. Γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα πετύχουν την επίτευξη μεγαλύτερη χρηματοδότηση Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Επιτροπή ε, εδώ συνειδητοποιούν ότι ε, θα πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό σε πολλούς από τους stakeholders ότι με τη μετατροπή σε μακροπεριοχές δεν θα έχουν περισσότερα κονδύλια αλλά το θέμα είναι ε, δεν είναι η δομή αλλά τα καθήκοντα. Δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη μόδα των μακροπεριοχών ή των ΕΟΕΣ γιατί τελικά τι θα κάνουμε. Θα εμπλέξουμε, ε, θα, θα προκαλέσουμε σύγχυση στους πολίτες. Οι μακροπεριοχές μας φαίνονται πολύ καλή πρωτοβουλία αν πρόκειται να μιλήσουμε για τη σύσταση δικτύων συμφερόντων. Η πρώτη μακροπεριφέρεια είναι η μακροπεριφέρεια τη Βαλτική, ε, για την οποία μιλάμε. μα φαίνεται λογικό να έχουμε μια τόσο τεράστια επικράτεια όπω η Βαλτική, όπου έχουμε πάρα πολύ μικρότητα, πυκνότητα πληθυσμού ε, με πολύ μεγάλε προκλήσει. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα συντονισμό μέσω του μοντέλου τη μακροπεριφέρεια. και ίσω αυτό θα ακολουθούσε περισσότερο τα προγράμματα του διεθνικού χαρακτήρα και όχι του διασυνοριακού χαρακτήρα και δεν αποκλείουμε ότι προγράμματα και διασυνοριακά αλλά και διαπεριφερειακά θα μπορούσαν να εκτελεστούν στο πλαίσιο μιας μακροπεριφέρειας. Γιατί όχι, αλλά ας, ε, ε, μην ε, προβαίνουμε στη δημιουργία τέτοιων μακροπεριφερειών έτσι ε, χωρίς ε, δεύτερη σκέψη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποια μακροπεριφερεια για το Δούνευ, παραδείγματος χάρη αλλά βλέπουμε και άλλες περιπτώσεις που πρώτα ήταν κοινότητες εργασίας μετά δημιούργησαν ευρωπαϊκούς ομίλους και τώρα θέλουν να αποκαλούνται μακροπεριφέρειες. Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω όταν μιλάμε για συνορική συνεργασία, οπότε δεν μιλάμε για αρμοδιότητε ούτε για νέα διοικητικά επίπεδα. Τα διοικητικά επίπεδα και τα πολιτικά είναι αυτά που είναι. Ή τι αρμοδιότητε τι έχουν αυτοί που του έχουν. Τα κράτη και κατόπιν ε, στο ιστορικά του κάθε κράτου ε, οι περιφέρειε ή οι δήμοι. Ανάλογα με το επίπεδο αποκέντρωση. Εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκά καθήκοντα, καθήκοντα που μπορούν να ανατεθούν. Ε, δεν μιλάμε για ανάθεση αρμοδιοτήτων, αλλά για καθήκοντα έτσι ώστε να γίνει καλύτερη ανάλυση γιατί υπάρχει καλύτερη γνώση στην περιοχή στα σύνορα και μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι stakeholder και μπορεί τελικά η εκτέλεση να είναι πιο κατάλληλη. Ε, και μιλώ για την εκτέλεση των προγραμμάτων των καθηκόντων. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη επίσης να αναλάβουν το ρόλο τους. Η επικουρικότητα δεν είναι ένα θέμα μόνο που αφορά τα ευρωπαϊκά όργανα, τους δήμους και τις περιφέρειες. Είναι και θέμα κρατών τελικά, γιατί όπως λέμε στα ισπανικά ε, τα κράτη είναι αυτά τελικά που ασκούν ε, την ε, εξουσία. Το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων το έχουν τα κράτη και θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που να δίνει λύσεις στις πολλαπλές ερωτήσεις που έχουν οι πολίτες. Χρειάζεται μια πραγματική συμμαχία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και διοικητικών επιπέδων, δηλαδή του Δήμου, της Περιφέρειας, του κράτους και της Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι μια απλή δήλωση σε ένα χαρτί, γιατί τελικά οι πολίτες είναι αντικείμενο αυτών των προγραμμάτων. Οποιοδήποτε μικρό σχέδιο, ακόμη και αν χρηματοστείτε με 4-5 εκατομμύρια ευρώ, τελικά θα έχει ένα δικαιούχο που είναι ένας ε, πολίτης που έχει ένα πρόβλημα σε κάποια παραμεθόριο περιοχή και με αυτή τη μικρή επένδυση η πιθανότατα θα έχουμε λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα για αυτό τον πολίτη και για την οικογένειά του. Δηλαδή πώς μπορεί να βρει δουλειά από την άλλη πλευρά των συνόρων, πώς ε, θα έχει ιατρική περίθελψη, κατάλληλη, ε, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να διασχίσει τα σύνορα πολλές φορές ή μπορεί να μάθει καλύτερα τη γλώσσα του γείτονα και να μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα στην αγορά εργασίας και πολλά άλλα πράγματα. Πολλά από αυτά τα προγράμματα κοστίζουν πάρα πολύ λίγο, αλλά χρειάζονται να υπάρχουν μικρά προγράμματα που να πτήσονται σε αυτό το επίπεδο, σε όλε τι παραμεθορίε περιοχέ, με την τάση να σκεφτόμαστε τα μεγάλα project, ε, τις μεγάλες πρωτοβουλίες ε, που υλοποιούνται από τις μακροπεριφέρειες. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα μικρά ε, προγράμματα να εγκαταλειφθούν, ενώ τελικά αυτά φτάνουν πιο κοντά στον πολίτη. Και επίσης θέλω να αναφερθώ και στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασυνοριακή και εδαφική συνεργασία επίσης γίνονται και στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το ότι εδώ μιλάμε για θεωρήσει για εξωτερικά σύνορα και για άλλου δυσκολίε. δυσκολίες. Υπάρχει εμπειρία που έχει επεκτηθεί για τη διασυνορική συνεργασία εδώ και δεκαετίες. Μπορούμε να ρωτήσουμε τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι η πρώτερη εμπειρία που έχουν για τη διασυνορική συνεργασία και σίγουρα θα μα απαντήσουν πολύ θετικά. Μιλάμε για ένα μοντέλο εξάσκηση για άλλε πολιτικέ, μεγαλύτερου ελληνικού και φυσικά πρέπει να ενταξούμε του πολίτε και σε μέσα όπως ο ΕΟΕΣ ε, έχουμε ε, βάλει κάποιες δυνατότητες για τη συμμετοχή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ένα κράτος που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρειάζεται για να συμμετάσχει να υπάρχει προϋπόθεση συμμετοχής άλλων δύο τουλάχιστον κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια πράγματα προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη και όσοι θέλουν να συζητήσουν το πρόγραμμα αυτών, το μέλλον αυτών των προγραμμάτων, όπω η κυρία Σέντσε Σμιθ, και να λάβουν υπόψη τη μελέτη για τη δυνατότητα να βελτιωθεί ο κανονισμό για του Ευρωπαϊκού Ομιλού Εδαφική Συνεργασία, Εμεί ε, μπορούμε να συμβάλλουμε. Έχουμε εξετάσει αυτά τα έγγραφα και πάρα πολλέ από τι ε, συνεισφορέ έχουν ληφθεί υπόψη και πρέπει να ευχαριστήσω και εσά, τα μέλη αυτή ε, τη επιτροπή που δείξατε ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε ότι ενδιαφέρεστε για το μέλλον τη εδαφική συνεργασία και που μα καλείτε τακτικά στις διάφορες περιφερειές και στους Δήμους, γιατί σας ε, βεβαιώνω κάθε φορά που σας κάνετε αυτό το εγχείρημα και εμείς αισθανόμαστε πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκίγερμο Ραμίρες. Και τώρα καλώ τον καθηγητή Σαρλ Ρίκ να μας παρουσιάσει και αυτό την δική του παρέμβαση. Καθηγητή Σαρλ Ρίκ Σαπί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πάντοτε χαρά και ευχαρίστηση να λαμβάνω το λόγο ενώπιον των Ευρωβουλευτών. Είμαι εδώ μαζί με την ε, συνάδελφο κυρία Σάντζεν Σμιθ, η οποία έχει δείξει το δυναμισμό που χρειάζεται πολλές φορές, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει όχι μόνο το παρελθόν και το παρόν της Ευρώπης αλλά και το μέλλον της ε, ως προς την περιφερειακή πολιτική. Κυρία Πρόεδρε, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει να μιλάνε για την περιφερειακή πολιτική ε, σε διάφορες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούμε πάντα να περάσουμε το, το μήνυμα αυτό της συνοχής θα προσπαθήσω να μιλήσω σε λίγα λεπτά. Ε, δύσκολο για ένα πανεπιστημιακό, ίσως για σας είναι πιο προφανές ως βουλευτές. Να πω ότι θα ήθελα να αναλύσω και να κάνω προτάσεις σχετικά με την διασυνοριακή ε, συνεργασία. Ο συνάδελφος Γιγέλμο Ραμύρες είναι υπεύθυνος για αυτή την ένωση των ε, εθωριακών περιοχών. Ο κύριος Λαμπέρς επίσης σε μια γερμανόφωνη περιοχή που ακολούθησε τον ε, Φανιστερρόη στην ε, Προεδρία. Γιατί μας ενδιαφέρουν τώρα οι παραμεθόρειες περιοχές. Θα έλεγα την προσωπική μου άποψη ο παππούς μου ήταν Βέλγος, ε, φλαμανδός ε, και δούλευε και αυτός ε, σε μια τέτοια μεθο... ζούσε σε μια μεθοριακή περιοχή και δούλευε σε μια διπλανή χώρα. Πήγαινε στη Νότια και στην Ελβετία ταυτόχρονα ε, και είχε αυτό το διασυνοριακό χαρακτήρα. Ε, θα σας ε, θυμίσω λοιπόν ποια είναι αυτά τα στοιχεία της διασυνοριακής συνεργασίας που μας, θα μας πάνε στο μέλλον. Οι μεθοριακές περιοχές πολύ περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες είναι αυτές που στην ιστορία καθόρισαν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Είναι ο καταλήτης, ε, ε, οι περιοχές αυτές που αποκάλυψαν ε, κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα, γιατί ουσιαστικά ενσωματώνουν τις ευρωπαϊκές ρίζες. Υπάρχει μια διαλεκτική λοιπόν σχέση. Εσείς ε, ως ευρωβουλευτές είστε οι πρώτοι που ανταποκρίνεστε σε τέτοια, μια τέτοια διαλεκτική. Υπάρχει μια μικροενσωμάτωση και ζυγίζω τους όρους μου ε, στις παραμεθόρες περιοχές ε, εν και σε σύγκριση με, την, με το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η μακροενσωμάτωση και ολοκλήρωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από ιδιότητες ε, συμπερίληψης, ε, αντιπροσώπευσης κτλ. Σε αυτά, ε, στις παραμεθόριες περιοχές, σε αυτούς τους χώρους της μικροολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης, που, γιατί λέγονται έτσι, θα σας πω κάποια παραδείγματα. έχουμε δημιουργήσει δεξαμένες ζωής, εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας, κινητικότητας, διαχείρισης εδάφους, πολιτισμού και διασκέδασης έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τους πληθυσμούς που ζουν εκεί. Έχω γράψει μία διατριβή ε, για το θέμα αυτό το 1978 και ανέφερα τους όρους ε, κόψιμο και ράψιμο. Εσείς μιλήσατε για κατακαιρματισμό, εγώ θα το έλεγα έτσι κόψιμο και ράψιμο. Και οι δείκτες που δείχνουν αυτό το κόψιμο δείχνουν ακριβώς και το ράψιμο. Αυτή η διαλεκτική λοιπόν μεταξύ μικρό και μάκρο ολοκλήρωσης. Τι γίνεται τώρα με το μέλλον. Ε, τα διάφορα στάθια πρέπει να γίνουν σεβαστά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 27 και στις 47 του Συμβουλίου του, της Ευρώπης. Πρέπει να έχετε λάβει το κείμενό μου. Ουσιαστικά προσπαθώ να συνοψίσω 30 χρόνια της ε, ζωής μου, παρελθόν, παρόν και μέλλον, ε, ως προς την διασυνοριακή συνεργασία. Υπάρχει μία λοιπόν αμοιβαία πληροφόρηση ε, που φτάνει μέχρι και την εκτίμηση του ε, γείτονος. Σε αυτούς τους ε, οργανισμούς και ελπίζω ότι όλοι εδώ είστε πεπισμένοι ότι το ότι τα μεγάλα ε, πολιτικά συστήματα είναι όλα δημοκρατικά, αυτά από τα οποία ε, εξαρτώμαστε, ο φεντεραλισμός κτλ. Περνάω από το ένα θέμα στο άλλο, λέει ο μιλητής. Όλα λοιπόν είναι δημοκρατικά και δείχνουν τρόπους λειτουργίας και εδαφικής οργάνωσης ε, που είναι διαφορετικά σε στη μία περιοχή και στην άλλη. Και οι παραμεθόρες περιοχές είναι ας πούμε ο συνδετικός ε, κρίκος, ε, είναι αποκεντρωμένες, ε, ομοσπο, ομοσπονδιοποιημένες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι. Είναι ο συνδετικός κρίκος που βοηθάει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Η δεύτερη διαπίστωση που έχετε ήδη αποδεχτεί στις 5 Ιουλίου του 2006 για την διασυνορική συνεργασία. Το πρόβλημα εν μέρη λύεται από την νομική προσωπικότητα των διασυνοριακών περιοχών. Μιλώ για τις ε, πράξεις των θεσμικών τους οργάνων. Έχει γίνει βέβαια πρώτο αυτό, θα το αναφέρω αργότερα. Δεύτερη διαπίστωση, σε όλες τι ε, συνοριακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πάντοτε το διαρκές ενδιαφέρον, όλα είναι διαρκή, δεν ξέρω, ίσως όχι πάντα. Όλα λοιπόν έχουν μια διάρκεια για να είναι και το ενδιαφέρον διαρκές. Θα πρέπει οι πολιτικές για τις περιοχές αυτές να είναι διαρκείς, ακόμα και αν αλλάζουν οι εξουσίες, οι πολιτικές. Ο ίστατος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ανθρώπινος συστός διασυνοριακών σχέσεων μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που υπάρχουν και στις δύο πλευρές των συνόρων. Μια άλλη διαπίστωση είναι το πρόβλημα των χρημάτων. Λίγες συνοριακές περιοχές έχουν τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς ε, προϋπολογισμούς που πραγματικά να έχουν ένα διασυνοριακό ε, χαρακτήρα. Το Interreg 4 από το 1991 ως τώρα έχει δώσει μια ευρωπαϊκή απάντηση ας πούμε στο πρόβλημα αυτό, το ειδικό πρόβλημα των παραμεθόρων περιοχών. την ειδική φύση της κάθε παραμεθόρειας, παραμεθόρειας περιοχής, κάτι που ξεχνάμε συχνά. Έτσι λοιπόν το θέμα αυτό του διασυνοριακού ε, προϋπολογισμού κατά κάποιο τρόπο επιλύεται επαρκώς. Πέμπτη διαπίστωση. Ε, θα γνωρίζετε ότι ε, πολλοί είναι οι βουλευτές που προέρχονται από παραμεθόριες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει να κάνει με τις οικονομικές ισορροπίες αυτών των περιοχών που εκδηλώνονται ε, στα πλαίσια της στέγασης, της εργασίας, ε, της αποσχόληση των μεταφορών και της ψηφιακής κοινωνίας η οποία και αυτή ε, επιζητά κάποιες συγκεκριμένες ισορροπίες. Κύριε Σάντζεσμιτ, και άλλοι Ευρωπαίοι βουλευτές που βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα, σας προτείνω ένα συγκεκριμένο καθεστώς, αν μου επιτρέπετε να το πω μάλιστα και πειραματικό, σε επίπεδο οικονομικό, φορολογικό, νομικό, κοινωνικό. Εδώ βέβαια μπορεί να υπάρχουν κάποιες, πληρο... δυσκολίες γιατί σε επίπεδο φορολογικό χρειάζεται μονοφωνία μεταξύ των χωρών όπως και σε κοινωνικό επίπεδο και γι' αυτό η ισορροπία πολλές φορές ε, μπορεί να διακυβεύεται από την έλλειψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε κάποιες περιπτώσεις και οι διασυνοριακές περιοχές ίσως θα ήταν μια απάντηση ίσως θα έφτανα μέχρι να προτείνω και μία ε, ας πούμε και ένα μαλάκωμα, μία χαλάρωση ε, των ευρωπαϊκών ε, οδηγιών, με κοιτάτε λίγο περίεργα βλέπω, που θα μας επέτρεπε να αναπτύξουμε καλύτερα σε αυτές τις παραμεθ... διασυνοριακές ευρωπαϊκές ε, περιοχές τους στόχους μας. Η τελευταία παρατήρησή μου έχει να κάνει πάλι με τις ανισορροπίες σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, φορολογικό, οικονομικό, νομικό επίπεδο. Επιμένουμε πολύ σε αυτά, ε, γιατί υπάρχουν τα πολιτιστικά και νοητικά σύνορα, όπως θα τα έλεγα. Είναι ξεκάθαρο ότι σε όλες τις παραμεθόρειες περιοχές της Ευρώπης υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, τα όρια του νου που πολλές φορές ενισχύονται και από την γλωσσική διαφορά μεταξύ των δύο κοινοτήτων και είναι ξεκάθαρο ότι θα ήταν καλό και εσείς ως ευρωβουλευτές ε, θα μπορούσατε να σπρώξετε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να υπάρχει μια διασυνοριακή ταυτότητα η οποία δεν θα αρνείται τις περιφερειακές ή εθνικές ταυτότητες που υπάρχουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πρόσθετη ιδιότητα, η οποία μέσα από τη συνέργεια θα μπορέσει να απαντήσει στα συνοριακά προβλήματα. Για να ολοκληρώσω την πρότασή μου, υπάρχει πάλι αυτή η διαλεκτική σχέση μεταξύ μικροολοκλήρωσης και μακροολοκλήρωσης. Ε, εσείς οι ευρωβουλευτές ε, από τις εκλογικές σας περιφέρειες, την περιοχή σας, ε, τις διάφορες διοικητικές και πολιτικές οντότητες από τις οποίες προέρχεστε, μπορεί να θεωρείτε ότι είναι ξεπερασμένη αυτή η διαλεκτική. Για να ανταποκριθούμε όμως στις συγκεκριμένες προκλήσεις των συνοριακών περιοχών που δείχνουν ότι είναι περιοχές οι οποίες χρειάζονται και πάλι να επανέλθει σε αυτές η ισορροπία ε, σε όλα τα επίπεδα ή χρειάζονται να αντιμετωπιστούν τα μοντέλα τους πολιτιστικά και μη που βάζουν ένα φρένο σε αυτήν την διασυνοριακή ε, συνεργασία χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ελπίζω να ήμουν συγκεκριμένο. Προσπάθησα να θίξω ε, εντάχει κάποια προβλήματα. Θα σας πω για παράδειγμα ότι η χρήση των νοσοκομείων από τη μία πλευρά και από την άλλη, η τροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα, ε, το πόσο αντιστοιχούν τα πτυχία, ε, η διασυνοριακή αστυνομία, ε, ειδικότερα για τη μάχη κατά των ναρκωτικών, εισιτήρια στις μεταφορές για διασυνοριακή μεταφορά κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Την ε, διάσκηση των συνόρων από τα ζώα. Ε, πολλές φορές γίνεται αυτό. Βλέπουμε τα ζώα να περνάνε 100 ε, χιλιόμετρα, πούμε, πιο πέρα να φτάνουν μέσα από τα σύνορα. Οι φορολογικοί κανόνες, κοινωνικές εισφορές, ε, ένα πολιτιστικό ε, διαβατήριο για να μπορεί κανείς να πηγαίνει ας πούμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μια τηλεφωνική συνεργασία για κάποια ε, χιλιόμετρα, ένα εγχειρίδιο διασυνοριακής ιστορίας. Όλα αυτά είναι λύσεις που εγώ από την πλευρά μου προτείνω, τολμώ να προτείνω και που θεωρώ ότι λύνουν αυτά τα προβλήματα διότι είναι ξεκάθαρο όσο ποτέ τουλάχιστον σε εσά τους βουλευτές ότι οι περιφέρειες αυτές αν φτάσουν σε αυτή τη μικρό ολοκλήρωση και ενσωμάτωση πραγματικά θα είναι η ενσάρκωση της Ευρωπαϊκής ε, Ενότητας στην οποία εγώ προσωπικά ονειρεύομαι και ελπίζω ότι όλοι μας ε, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα θα καταφέρουμε να πετύχουμε. Γιατί λοιπόν ε, να μην φανταστούμε μια μέρα όπου θα έχουμε ευρωπαϊκές ε, διασυνοριακές ε, περιοχές οι οποίες θα εκλέγουν και δικούς τους βουλευτές. Φτάνω πολύ μακριά όμως αυτό είναι και αυτό μια πρόταση και για να καταλήξω να πω ότι παραμεθόρες περιοχές είναι ο καταλήτης για την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, κύριοι Ευρωβουλευτές και συνάδελφοι. Uh, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι τέθησαν πολύ σημαντικά ε, ζητήματα και από τους δύο ε, καλυσμένους ομιλητές μας και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε ε, αυτή την έκθεση το Μάρτιο και θα την έχουμε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Επομένως, έχουμε την ευκαιρία, ίσως την τελευταία ευκαιρία, να επηρεάσουμε ε, την κατεύθυνση των εργασιών για την εδαφική συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των κανονισμών που θα παρουσιαστούν στα μέσα του επόμενου χρόνου. Και επομένως αυτή η έκθεση δεν πρέπει να είναι μόνο μια γενική έκθεση για τη σημασία της διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, αλλά θα πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένα αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πού θα θέλαμε να προχωρήσει η ε, εδαφική συνεργασία. Σας καλώ λοιπόν να συνεργαστείτε στενά με την κυρία Σάντσε Σμιτ έτσι ώστε να έχουμε την έκθεση ε, που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να διαπορφώσουμε το μέλλον της εδαφικής συνεργασίας. Σας καλώ λοιπόν να ανοίξουμε τη συζήτηση και η κυρία Μαλέσκου είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτό το έγγραφο και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ε, καλεσμένους που ε, μοιράστηκαν μαζί μας κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες. Ε, σε γενικές γραμμές είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε και προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις και λύσεις. εάν αναφερόμαστε στη μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακή διεθνική και διαπεριφερειακής συνεργασίας και θέλουμε να είναι πετυχημένοι, θα πρέπει να δώσουμε στις τοπικές και περιφερειακέ αρχές την εξουσία που χρειάζονται. Πρέπει να αρθούμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα διαπεριφερειακά ε, προγράμματα, ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην διαπεριφερειακή συνεργασία, ιδιαίτερα μετά το 2013, στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Για τη διακυβέρνηση τώρα και την σημασία της ε, εδαφικής ε, διακυβέρνησης. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για την πραγματική εφαρμογή της εδαφικής συνοχής. οι περιφέρειες έχουν ένα δυναμικό το οποίο δεν χρησιμοποιείται σωστά και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό σημείο σύγκλησης των ε, κοινοτικών πολιτικών. Για να παγιωθούν οι περιφερειακές πολιτικές θα πρέπει να προωθήσουμε την διαπεριφερειακή ε, συνεργασία και να έχουμε ανταλλαγή ε, εμπειριών. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε ε, ανοιχτοί σε πιθανούς εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία. Ενθαρρύνοντας λοιπόν τις επιχειρήσεις και τους ομίλους έρευνας να συμμετάσχουν. Είναι σημαντικό λοιπόν να δοθεί ευκαιρία στους ιδιωτικούς εταίρους να γίνουν ε, πλήρη μέλη σε αυτά τα προγράμματα. Επίσης, χαιρετίζουμε την αναφορά της εισηγήτριας στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας, ο οποίος ενισχύει αυτή τη συνεργασία και πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από τα κράτη-μέλη για τα συστήματα διασυνοριακής διακυβέρνησης, καθώς και για την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Καλούμε τα κράτη-μέλη που δεν χρησιμοποιούν ακόμα αυτόν τον όμιλο να υιοθετήσουν τις απαραίτητες διατάξεις για την δημιουργία τέτοιων ομίλων για την εδαφική συνεργασία. Και στην δική μου ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας καλώ την κυβέρνησή μου να το κάνει. Για τα επιχειρησιακά ε, προγράμματα ε, υπάρχει μια έλλειψη πολιτικής βούληψης σε εθνικό επίπεδο και υπάρχει μια μικρή συμμετοχή των διαπεριφερειακών πολιτικών. Αυτό είναι το πρόβλημα της μη συμμετοχής των εθνικών και τοπικών ε, αρχών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τη συμπερίληψη του προγράμματος Εράσμους για τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις στην διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία με την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς για τις ε, πληροφορίες και για την έκθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας, η οποία είναι πλήρης. Υπάρχουν κάποια κεντρικά σημεία που θίγονται και αυτά ίσως μπορέσουμε στην Επιτροπή να τα θίξουμε. Αλλά θα εκμεταλλευτεί την παρουσία των εμπειρογνωμόνων για να θέσω κάποια ερωτήματα για την διασυνοριακή συνεργασία. Κατάλαβα, αλλά τελικά ποια είναι τα σημεία κλειδιά, τα απτά σημεία κλειδιά τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να προσαρμόσουμε. Και μιλάω και για τα σύνορα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη συνεργασία σε αυτές τις ε, περιοχές. Ε, πόσο κοντά μπορεί να είμαστε, πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε, αν είμαστε ευέλικτοι ή όχι. Και έχω και άλλο ένα ερώτημα τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Δεν πρέπει σε συγκεκριμένες ε, χώρες να ε, έρχονται περισσότερα από τις περιφέρειες. Άκουσα πολλά, αλλά ε, δεν υπάρχει τόσο μεγάλος ενθουσιασμός όπως με την Ευρώπη 2020. Έχουμε ακούσει για προγράμματα σημαίες και τα λοιπά, αλλά για το 2007-2013 την προηγούμενη προσαρμογή τα εξωτερικά σύνορα της χώρας κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε δει πώς, πώς θα γίνει ε, πρέπει λοιπόν να πω σύντομα ότι για τα εξωτερικά σύνορα ότι στην έκθεση δεν αναφέρονται αρκετά επαρκώς αυτά που θέλουμε. Υπάρχουν ζητήματα χωριστά που έχουν τεθεί ως ερώτημα για τα προγράμματα γυπνίασης. και ίσως πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτή η πολιτική γυμνίασης είναι κάτι που πραγματικά με ανησυχεί. Τι γίνεται με τα εξωτερικά σύνορα. Έχω την αίσθηση ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στην, στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι στα εξωτερικά. Ίσως βέβαια κανείς ε, να πρέπει να πει ότι τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία. Όμως ε, μέσα από αυτό το έγγραφο εργασίας ίσως θα ήταν καλό ε, να δούμε αυτά τα θέματα και μέσα από το τελικό πρόγραμμα, ε, έγγραφο της κυρίας Σάντσες. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Σάντσες ε, για αυτή τη βάση που μας δίνει για περαιτέρω συζητήσεις και ένα έγγραφο εργασία για αυτή την Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα που έχουν σημασία στις συνοριακές περιοχές. Επίσης, να ευχαριστήσω τους ομιλητές ε, σήμερα που μας έδωσαν μια άλλη άποψη για την προβληματική, ειδικότερα για την εργασία σε διασυνοριακές περιοχές. Ε, για τον κύριο Ραμίος ειδικά που μίλησε για τις μακροπεριφέρειες. Βλέπω ότι μιλήσατε από ψυχής, από καρδιάς ε, και τελικά οι μακροπεριφέρειες είναι κάτι διαφορετικό από τις διασυνοριακές περιοχές που λέγαμε εμείς. Μια κοινή λοιπόν στρατηγική ε, δεν είναι αυτό που θα ε, αντικαταστήσει την άμεση εργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις διασυνοριακές περιοχές. Δεν είναι μια εναλλακτική, είναι μια προσθήκη θα λέγαμε στην ευρύτερη στρατηγική. Ε, σκέφτομαι λοιπόν ότι στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των συνοριακών περιοχών με πολύ περισσότερη εργασία. Τώρα, πώς θα διαρθρωθούν τα προγράμματα Έχουμε το Interreg 4 για παράδειγμα, το οποίο έχει βοηθήσει στην εκπλήρωση τέτοιων προγραμμάτων. Εγώ είμαι, στο, είμαι από το Άχεν. Εκεί έχουμε μια καλή συνεργασία διασυνοριακή και σκέφτομαι ότι παρόλο που υπάρχουν οι διάφορες ε, εθνικές διατάξεις που δυσκολεύουν τα πράγματα, ε, τα προγράμματα λειτουργούν καλά και ε, πραγματικά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε που μπορέσαμε πρακτικά να έχουμε εμπειρία ε, σε μια τέτοια διοσιονοριακή συνεργασία έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τις περιοχές αυτές και να βρούμε τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες μέσα από τους διασυνοριακούς μηχανισμούς ελέγχου θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Τα σύνορα λοιπόν έχουν αρθεί σε πολλές περιοχές, όμως υπάρχουν και πολιτικές όπου ε, ακόμα ισχύουν και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις ε, παραμεθόρες περιοχές. Ας πούμε η υγεία, τηλεφωνικές, τηλεφωνικά τέλη, μεταφορές κτλ. Η, η προστασία από καταστροφές, από πυρκαγιές. Μπορεί να έχουμε κάποιον ο οποίος βρίσκεται κοντά στα σύνορα και να απειλείται από τέτοια πράγματα. Ε, αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να απλουστεύσουμε στο μέλλον το πιο σημαντικό θεωρώ είναι ότι μέσα από το πρόγραμμα Interreg και άλλες τέτοιες συνεργασίες μπορούμε να προχωρήσουμε. Όταν σκέφτεται κανείς το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής και μιλάει γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ο στόχος 1 και 2 θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ε, παραμεθόρες περιοχές όλο και περισσότερο. Ε, ας πούμε, ε, υπήρχαν περιπτώσεις που είχαμε κατασκευή δρόμων όπου ήταν μεγάλες οι δυσκολίες ε, που αντιμετωπίστηκαν και οι διαφορετικοί κανονισμοί ε, που δυσκόλευαν την κατάσταση για την χρήση των ιδίων κονδυλίων κτλ. Ελπίζω λοιπόν ότι στο μέλλον το χρηματοδοτικά μέτρα μέσα του Ίντερεγ θα, θα πρέπει να προσαρμοστούν και σε αυτά τα δεκομένα, δεδομένα. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ, Ρίκα Μάνεν. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό έργο της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε και εμείς να συζητούμε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα πάντω ε, να μιλήσω για τα εξωτερικά σύνορα και μπορώ να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Βανίστη ότι θα πρέπει να επιμείνουμε επί του θέματος αυτού και να κάνουμε μια συζήτηση βάθο γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στα προγράμματα για τα εξωτικά σύνορα. Εγώ προέρχομαι από την Ανατολική Φιλονδία, κοντά στα ρωσικά σύνορα και ξέρω ότι τα προγράμματα δεν λειτουργούν πολύ καλά. Υπάρχει πάρα πολύ δυναμική σε αυτή την περιφέρεια, αλλά δεν μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε πλήρως. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με αυτό το πρόγραμμα ε, Interact που δεν λειτουργήσε καλά είναι το πρώτο. Δεύτερον, ε, η Ρωσία πρέπει να θεωρηθεί μία αναπτυσσόμενη χώρα, όμως αυτό δεν το βλέπουν ε, πολύ καλά από τη ρωσική πλευρά και το ENPI, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας Κεντρικής Σχέσης θα πρέπει να ενταχθεί στην πολιτική συνοχή. Εγώ είμαι υπέρ αυτής ε, της ε, μεταφοράς και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και με την Κομισιόν γιατί στην πολιτική συνοχή σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο λειτουργικοί από ότι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και η κυρία ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, καταρχήν ε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και συμφωνώ με τον κύριο Βανίλιστελ Δεν ε, λέγονται αρκετά για τα εξωτερικά σύνορα. Από ό,τι φαίνεται, το ίδιο το θέμα παραγωνίζεται καθώς ε, εμείς έχουμε εξωτερικό σύνορο μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας. Ε, είναι ε, πάρα πολύ διαφορετική συνεργασία και η δυναμική και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες διαφορές γιατί έχουμε εμείς ε, ως ε, νέο κράτος μέλος μικρότερη εμπειρία. Και η συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα πολλές φορές είναι μέχρι και αδύνατη και θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, πρώτερη δήλωση ότι στις παραμεθόριες περιοχές ε, υπάρχει διαφυγή των νέων. Νομίζω ότι αυτή η φυγή της ε, νέας γενιάς Αυτή τη φυγή τη βλέπουμε κυρίως ε, σε παραμεθωρείς περιοχές που είναι κοντά στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παραδείγματος χάρη ένας από τους παράγοντες είναι η ιατρική περίθαλψη. Αναφέρθηκε και αυτό από τον κύριο καθηγητή. Αν δείτε τι συμβαίνει στην Ουκρανία έχουν εντελώς διαφορετικά συστήματα και νομοθεσία. Ναι για τους Ουκρανούς θα μπορούσε να είναι εξαιρετική λύση, αλλά για μας θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σηκώσουμε το κόστος. Έτσι λοιπόν, η δική μου άποψη θα ήταν να σκεφτούμε καλύτερα όλο αυτό το ζήτημα όταν αναφερόμαστε στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις σχετικές παραμεθόρες περιοχές, γιατί εκεί η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτά που προτείνονται για άλλα σύνορα δεν μπορούν να εφαρμοστούν ε, και στα εξωτερικά σύνορα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να πάρω εγώ το λόγο, γιατί πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και πολύ σημαντική η έκθεση και θα πρέπει να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τη μελλοντική πολιτική. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτών που μπορούμε να δούμε από την πολιτική συνοχή ήδη, η εστίαση μετά το 2013 θα είναι στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής και η σχέση μεταξύ ε, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διασυνοριακή ε, πολιτική όπως την ξέρουμε και όπως φαίνεται στις παρουσιάσεις των μιλητών, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά ταμεία με έναν τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και γι' αυτό θα πρέπει να καταργηθούν όλα τα εφιστάμενα εμπόδια στην ενιαία αγορά που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν εάν μπορούσε η κυρία Σάντσες να ε, εισάγει αυτή την προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε δηλαδή ότι θα υπάρχει μια νέα προσέγγιση στην ενιαία αγορά για να ευξήσουμε την αποτελεσματικότητα και να μιλήσουμε και για τη συνεργασία της αστυνομίας, των κοινωνικών υπηρεσιών κτλ. έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην διασυνοριακή συνεργασία. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς για ορισμένα μερικά πράγματα στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Λαμπέρ, για παράδειγμα το πρόβλημα των 150 χιλιόμετρων, ένα πρόβλημα που όλοι ξέρουμε. Υπάρχει το θέμα της διαφοροποίησης ανάμεσα σε διάφορες περιοχές των κρατών μελών κάτι το οποίο επίσης ε, δημιουργεί προβλήματα. Επίσης υπάρχει το θέμα της επιλεξιμότητας μέσα στους ε, κανονισμούς και για το κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες των παραμεθόριων περιοχών. Πρέπει επίσης να προσαρμόσουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα που στο μέλλον θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει λοιπόν να τα προσαρμόσουμε στις ανάγκες της διασυνοριακής συνεργασίας και υπάρχουν και άλλα θέματα που αναφέρθηκαν από τον κύριο Λαμπέχ. Για παράδειγμα, για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονία και τερικής Σχέσης, πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το υφιστάμενο σύστημα και υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω και τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν προετοιμάσουμε αυτή την έκθεση. Γιατί είναι πραγματικά η ευκαιρία μας να έχουμε μια ε, επίπτωση, μια, έναν αντίκτυπο στην ε, μελλοντική πολιτική. Σε αυτό το στάδιο δεν μιλάμε για τη χρηματοδότηση, γιατί αυτό γνωρίζουμε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα και θα εξαρτηθεί από τις ε, γενικές αποφάσεις για την δημοσιονομική προοπτική. Όμως μπορούμε και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να εξετάσουμε την ε, πιθανότητα να αυξήσουμε την χρηματοδότηση για την, κοινωνική, για την πολιτική κοινωνική συνοχής γιατί είναι σαφής εδώ η ευρωπαϊκή προστιθέμενη ε, αξία. Και μία αύξηση 15% ε, θα ήταν ένα πολύ μικρό τμήμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής δεν είναι πολύ υψηλότερο από το ποσοστό που έχουμε σήμερα, όμως θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ε, πολιτικής. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σάντσες, εάν έχει άλλα σχόλια. Δεν θα πάρουμε αποφάσεις σήμερα. Θα επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση ε, για το προσχέδιο της έκθεσης στα τέλη του Ιανουαρίου, εάν συμφωνείτε κυρία Σάντσες. Σας δίνω λοιπόν το λόγο και μετά θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία, οπότε μην φύγετε από την αίθουσα, παρακαλώ συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Έχετε δίκιο με αυτήν την έκθεση και τη στρατηγική που θα προτείνουμε. Έχουμε μια ευκαιρία να επηρεάσουμε τις μελλοντικές αποφάσεις για αυτόν τον στόχο που είναι μέρος της ε, πολιτικής ε, συνοχής. Κατά, τις, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και της ανταλλαγής απόψεων που είχαμε, δεν αμφιβάλλουμε σίγουρα για την προστιθέμενη αξία της ε, πολιτικής για την εδαφική συνεργασία, τόσο και οι βουλευτές που έχουν αυτή την εμπειρία από τις περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται, όσο και οι ομιλητές, μας παρουσίασαν ότι έχουμε αρκετά προβλήματα, τα εμπόδια, όμως πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Συζητήσαμε για τις εταιρικές σχέσεις με τις τοπικές αρχές, ε, για την εφαρμογή. Όσον αφορά τα υφιστάμενα μέσα, είναι ε, αποτελεσματικά, ίσως όμως δεν χρησιμοποιούνται στο μέγιστο βαθμό. Είπατε ότι η μελλοντική πολιτική θα υπογραμμίσει κυρίως την αποτελεσματικότητα. Έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για αυτή την αποτελεσματικότητα. Πρέπει λοιπόν να τη βελτιώσουμε περαιτέρω. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή κάποιες συζητήσεις για τη χρηματοδότηση της χρηματοδοτήσεις μέσω της ε, διάρθρωσης, μέσω της δομής που έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιούμε για αυτή την πολιτική. Το θέμα που τίθεται τώρα είναι ποιο θα είναι το ποσό και ποια θα είναι και η κατανομή ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές και πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε οπωσδήποτε την πολιτική για την εδαφική συνεργασία. Άκουσα και αυτά που είπατε για τις μακροπεριφέρειες. Θα έχουμε σίγουρα μία συζήτηση επί της ουσίας για αυτή την ε, πολιτική είμαι πεπισμένη ότι δεν πρέπει να είναι μια πολιτική που θα επιβληθεί, θα πρέπει απλά να είναι ένα επιπλέον ε, ε, μέσο για κάποιες περιφέρειες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να δούμε την υφεστάμενη νομοθεσία και αυτή που θα μπορούμε να αναπτύξουμε, πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Είμαι ανοιχτή σε όλες τις συνεισφορές σας. Άκουσα τις προβληματικές που ετέθησαν θα τις λάβω υπόψη μου στην έκθεσή μου. Όπως είπατε και εσεί έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι το Μάρτιο και χαίρομαι ε, γιατί δεν πρέπει να προετοιμαστεί βιαστικά αυτή η έκθεση. Πρέπει να έχουμε όλο το χρόνο για τον απαραίτητο προβληματισμό. Σας ευχαριστώ. Και πάλι Ευχαριστώ τον κύριο Γκυγέρμο Ραμύρες και τον καθηγητή ε, Ρίκ για τις συνεισφυρές τους. Σας ευχαριστούμε. And thank you very much, ε, Και ε, σας ευχαριστούμε Μαρή Τεγρές. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Love those last minute lists. Uh, I would like to check the... Να ελέγξουμε τις ε, κάρτες για να κάνουμε μια δοκιμή, για να δούμε αν ε, λειτουργούν οι κάρτες της ψηφοφορίας. Μπορείτε να ανάψετε το σύστημα. So the vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Uh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 So here, here they are. No, it's, it's now 37 we have. You are ready, you tell me. Όταν είστε έτοιμοι μπορούμε να ξεκινήσουμε, να με ενημερώσετε. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με το σημείο 11 της ημέρας της διάταξης ε, και πέρα από αυτό μέτρες της πρόοδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, όπως ξέρετε. Έχουμε πάνω από 90 τροπολογίες. Ήταν ε, πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και μπορώ να πω ότι είναι επώδυνη διαδικασία. Πολλές φορές έχουμε λοιπόν συμφωνήσει επί 7 συμβιβασμών σε δύο σύνολα 7 συμβιβαστικών προτάσεων, διορθώνει ομιλήτρια, και πιθανότητα θα καθυστερήσουμε λίγο περισσότερο κατά τη διάρκεια της πληροφορία για να είμαστε σίγουροι ότι θα τα κάνουμε σωστά. Ας ξεκινήσουμε με την τροπολογία περιθμών 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλιστα, εγκρίνεται. Ας περάσουμε στον συμβασμό υπαριθμών 1 από τον εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Κανείς δεν επιμένει να ελέγξουμε. Λοιπόν, να σε ελέγξουμε και να δούμε για τη συμβιβαστική πρόταση 1 από τον συγγητή. Πέρα τη προφορίες. Απορρίπτεται. 24 κατά, 14 υπέρ. Ας περάσουμε τώρα στη συμβιβαστική πρόταση ΕΛΚ Φιλελεύθερη Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται με σαφήνεια. Ας περάσουμε στη συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας περάσουμε στο συμβασμό 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α περάσουμε στη συμβαστική πρόταση 3 από τις πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη τροπολογία 22. Υπέρ για την 22. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας περάσουμε στη συμβαστική πρόταση 4 από τον συγητή υπέρ. Δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, ε, το πρώτο μέρος για το συμβασμό 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας περάσουμε στο συμβασμό 4. Πολιτικές ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας περάσουμε στην τροπολογία περθνών 33. 36 διορθώνει ομιλήτρια. μιλήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και να ελέγξουμε. Για την τροπολογία 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 κατά 17 υπέρ. Ας περάσουμε στο συμβιβασμό 5 από τον εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπαριθμών 5 συμβιβασμός από τις πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός υπερθών 6. Από τον εισηγητή. Υπέρ. Για το συμβασμό 6. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 6 από τις πολιτικές ομάδες. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνδεσμός υπεριθμών 7, όπου και αν είναι. Ελπίζω να το βρήκατε από τον εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός υπερθυμών 7 από πολιτικές ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Τροπολογία υπερθυμών 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται κατά την άποψή μας περάσουμε στην 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ας περάσουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας και έχουμε 36 υπέρ 3 κατά ο κύριος Σουσπάσκης ζητά το λόγο. Δεν έχετε την κάρτα σας. I'm sorry, I can't. We can't hear, could you just speak? I'm sorry, I'm just, yeah. Uh, sorry, bet aš neturiu kartelės su savimi. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω φέρει μαζί μου την κάρτα μου σήμερα. Δεν το είπατε νωρίτερα όμως. Ε, θα σας μετρήσουμε για τις επόμενες ψηφοφορίες. Τώρα για αυτήν εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Φανίστη Λιρόι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα συγχαρώ για την ε, ψηφοφορία. Έχω μια ερώτηση για τον ε, εισηγητή. Ε, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα που βγαίνει από την ψηφοφορία. Να εκφραστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, θα το έλεγα κι εγώ κύριε συνάδελφε. Δεν σχετίζω πλέον το όνομά μου με αυτή την έκθεση και λυπάμαι γι' αυτό από τη στιγμή που οι συμβιβαστικές ε, τροπολογίες είναι ε, ε, τροπολογίες που πηγαίνουν ενάντια στο πνεύμα και τη δυναμική που θεωρούσα ότι θα έπρεπε αυτή η Επιτροπή να δώσει. Άρα αποσύρω το όνομά μου από αυτή τη γνωμοδότηση στην έκθεση. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος που θέλει να λάβει το λόγο. διαδικαστικό, παρακαλώ. Δικό σας ο λόγος. Λάθος, θα ήθελα να ξέρει το σώμα ότι εγώ τελικά έχω καταψηφίσει την έκθεση για την οποία μιλάμε. Άρα στις αρνητικές ψήφους σας παρακαλώ να προσθέσετε και τη δικιά μου. Θα τη διορθώσω και αργότερα. Ευχαριστώ. That's done. Έγινε. Κάποια άλλα σχόλια για αυτό το θέμα η διαδικασία. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι, δεν έχω την κάρτα μου μαζί. Θα μου την φέρουν, εάν πρέπει να τη χρησιμοποιήσω για αυτή την ψηφοφορία. Θα τη ζητήσω να μου τη φέρουν. Άρα έχουμε τρία άτομα που δεν έχουν κάρτα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να προσθεθούν οι ψήφοι αυτών των τριών ατόμων στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Από ό,τι κατάλαβε, η μία ψήφος είναι κατά. Εσείς κύριε Ρισπάσκη είστε υπέρ και εσείς. κύριε Χέιερ, είστε υπέρ ή κατά. Υπέρ. Αν δεν έχετε αντίρρηση, λοιπόν, να τις προσμετρήσουμε στην τελική ψηφοφορία. Και τώρα σχετικά με τη διαδικασία για την κατάσταση που έχει προκύψει. Δηλαδή, ε, αποσύρει ο εισηγητή το όνομά του από την έκθεση. Δυστυχώ, η μόνη λύση από ό,τι κατανοώ που έχουμε νομικά στη διάθεσή μας είναι να βάλουμε το όνομα του Προέδρου της Επιτροπής ε, στην έκθεση και να βάλουμε ένα επεξηγηματικό σημείωμα. Και είναι ο μόνος τρόπος που βγαίνουμε από αυτή τη δύσκολη θέση αν Κανείς δεν θέλει να πει κάτι άλλο σχετικά. Να κλείσουμε με αυτό το σημείο της σας διάταξης και να περάσουμε στο σημείο 12. Ε, γνωμοδότηση κυρίου Μποστινάρου για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μαύρη Θάλασσα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι? Ξεκινούμε λοιπόν με την ε, συμβαστική λύση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξεκάθαρα απορρίπτεται. Συμβαστική λύση 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 3. Να τη βρω λίγο. Υπέρ. 3. Λαμπέρ 3. Συμβαστική λύση 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε λίγο για την τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση. 20 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε λίγο με τα μέλη. Οι συνάδελφοι που δεν έχουν κάρτα, κύριε Σουσπάσκη, είναι κατά. 21 κατά, 21 υπέρ. κατά. 22 κατά. Όσοι θέλαν το υπέρ, Δυστυχώ απορρίπτεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν ξέρω, ας ελέγξουμε για την τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Συμβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 39. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 44. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 15 κατά, ξεκάθαρα εγκρίνεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορική υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν όλοι. Κλείνουμε την ψηφοφορία. 37 υπέρ, ένας κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια τον εισηγητή, τον κύριο Ποστινάρου. Για την τελική ψηφοφορία τώρα οι συνάδελφοι, οι τρεις συνάδελφοι ψήφισαν υπέρ, αυτοί που δεν είχαν κάρτες. Ναι. Ευχαριστούμε. Σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, η, έκθεση της κυρίας Φιλής Χάκεβα και Σουσάνοβα, εφαρμογή της οδηγίας 2006 123 ΕΚΑ υπηρεσιών. Πάμε στη συμβασική λύση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Compromise 2. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Έχουμε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές απο, ε, εγκρίνεται. Τμήμα 2, υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται Όμω θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. 27 κατά, επομένως απορρίπτεται. 14 υπέρ. Συμβασμός 3 υπέρ. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Συγγνώμη, διορθώνει ομιλήτρια. Τροπολογία 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ε, ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 2 κατά και μία αποχή και οι τρεις συναδελφοί είναι που δεν έχουν τις κάρτες τους είναι υπέρ. Ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Και περνάμε στο σημείο 14 βιομηχανική πολιτική, ε, γνωμοδότηση του Φρανσέσκο Ντεάντζελης. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 22 υπέρ, 20 κατά, επόμενος εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρουμε, θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 23 υπέρ, 20 κατά. Θα ήθελε κάποιος να προσθέσει την ψήφο του. Όχι. Εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θα το ελέγξουμε. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας 27 υπέρ 16 κατά. Κρίμα που δεν τον παρατήρησαμε πριν. Τροπολογία 17 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά δεν ξέρω, θα ψηφίσουμε λοιπόν για την 21 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας 22 υπέρ, 20 κατά. Όσοι δεν έχουν κάρτα θα ήθελαν να ψηφίσουν. Όχι, επομένως εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε. Εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 23. Πέρας της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. Τροπολογία 24, λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. ψηφίζεται πέρα τη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 21 κατά. Πώ θα μπορούσα να είμαι σίγουρη. τροπολογία 25 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται Συμβασμός 3 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 31. Υπέρ, κατά αποχές πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω πρέπει να το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 31 πέρας της ψηφοφορίας 28 υπέρ 15 κατά τροπολογία 33 Έχουμε μια προφορική τροπολογία από τον κύριο Διάντζελης. Είναι κανείς κατά, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 5, 4 ε, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Καταπίπτει. Δεν έχει εγκριθεί το 35. Επομένως δεν καταπίπτει το, η 36. Πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε για την 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 21 κατά. Θέλει κάποιος να προσθέσει τη ψήφο του. Εγκρίνεται τότε. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Ελέγχουμε για την 41 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας 25 υπέρ 18 κατά. Εγκρίνεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 27 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Ε, υπάρχει κάποιος, ε, κάποια αντίδραση στην προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψήφος, ηλεκτρονική, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 40 υπέρ, 1 κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια για τον κύριο Ντάντζελης. Και τώρα... Dear colleagues, I have a proposal. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια πρόταση, γιατί έχουμε κερδίσει μισή ώρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα τις ιδρύσεις των συντονιστών και μετά ε, στις 5 και 4 έχουμε τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των συλλόγων του Κλεισί Σουμποά. Μήπως οι συντονιστές θα μπορούσαν ε, να μην αποσπώνται από τους ε, διπλανούς τους. Κάνα μόλις μία πρόταση για τους συντονιστές. Καθώς τώρα έχουμε μισή ώρα χρόνο, Μήπω θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συνάντηση των συντονιστών τώρα ή θέλετε να κάνετε διάλειμμα. No. So, dear members of the Regi Committee... Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, όποιος δεν συμμετέχει στη συνάντηση των συντονιστών πρέπει τώρα να φύγει, να εγκαταλείψει την αίθουσα για μισή ώρα, να επανέλθετε στις 5 και 4 και να ξεκινήσουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Δύο λεπτά δίνω. Όλοι όσοι δεν συμμετέχουν στις συνεδρίες των συντονιστών παρακαλώ να καταλήψουν την αίθουσα. Και να επανέλθετε στις 5 και 4.